Πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχει σφυράκι, τι γίνεται. Λοιπόν, πολύ καλά. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας για σήμερα το απόγευμα. Ησυχία. Vamos Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας την απογευματινή. Προανήγγυλαν ότι δημιουργήθηκε ένα μικρό κενό εξουσίας, προσωρινό κενό εξουσίας, σαν συνέπεια των, του αποτελέσματος των εκλογών στη Γερμανία. Στους φακέλους σας έχετε στη διάθεσή σας ένα σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ελπίζω ότι μπορεί να εγκριθεί από πλευρά σας. Τώρα όσον αφορά αυτό το σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω για τους ίδιους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι στην Προεδρία και προεδρεύω αυτή τη στιγμή, θα έχουμε την έκθεση για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας αύριο το απόγευμα, ώστε ο εισηγητής Έλμαρ Μπρόκ να είναι παρόν και να μπορέσει να συνοδεύσει τις εργασίες μας. Δεν έχω άλλες παρατηρήσεις να κάνω σε σχέση με την ημερήσια διάταξη. Αν συμφωνείτε, περνάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 28 Αυγούστου. Ως ήθιστε, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις από πλευρά των μελών που θα κατατεθούν στη γραμματεία θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται αυτά τα πρακτικά. Και περνάμε λοιπόν στο σημείο 4 που είναι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΣΕΑΝ. Γνωρίζετε ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ήταν η 10η Σεπτεμβρίου ήδη. Οι συνάδελφοι θα βρουν στους φακέλους τους ε, τα όσα έχουν κατατεθεί είναι 112 τροπολογίες συνολικά έχουμε και την παρουσία του εισηγητή ανάμεσά μας, του κυρίου Μπιούτι Κόφερ. Τον ευχαριστούμε για την επιμέλεια που είχε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μετά από τις εκλογές που διεξήχθησαν εχθές στη χώρα του. Κύριε εισηγητά, λοιπόν, έχετε αμέσω τον λόγο για να μας κάνετε λόγο για το πώς έχει η έκθεσή σας αυτή τη στιγμή και τι θα κάνετε με αυτές τις 112 τροπολογίες που εξετάζονται. Κύριε εισηγητά, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από τις ε, εκλογές και τον θόρυβο που έγινε χαιρόμαστε που ήρθαμε στις Βρυξέλλες να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό ήθελα έτσι σύντομα να σας πω πως έχουν τα πράγματα. Εγώ βλέπω εδώ πέρα 112 τροπολογίες για τις οποίες ευχαριστώ τους συναδέλφους, τις οποίες είδα λεπτομερώς. Πρότεινα συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες ελπίζω να συζητηθούν στο επόμενο Στρασβούργο εάν πάνε έτσι τα πράγματα όπως ελπίζω, τότε οι μισές από τις ε, τροπολογίες θα αντικατασταθούν από τις συμβιβαστικές και με το σχέδιο καταλόγου ψηφοφοριών θεωρώ πως έχουμε το πολύ 20 ε, τροπολογίες που θα είναι επίμαχες. Βλέπω λοιπόν αρκετά μεγάλη συνένεση και νομίζω πως θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπιντικόφερ. Θα δώσω τον λόγο πρώτα στους κοιόδης εισηγητές των διαφορετικών πολιτικών ομάδων για να έχουμε μια συζήτηση με τα, με τα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Γέγκλε πρώτα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Μπουτικόφερ. Εντάξει, εμείς τα πήγαμε κάπως πιο καλά στις εκλογές, αλλά η δουλειά μας εδώ πέρα συνεχίζεται. Για μένα τρία πράγματα είναι σημαντικά και ένα τέταρτο που συνοψίζει τα πράγματα. Οι χώρες ε, του ΑΖΙΑΝ είναι οικονομικοί εταίροι. Είναι εταίροι στον τομέα της ασφαλείας και επίσης ε, στο κοινοβουλευτικό επίπεδο και το τέταρτο και για μένα αποφασιστικό όλα αυτά που είδαμε και επεξεργαστήκαμε αφορούν αποφασιστικούς τομείς. Γι' αυτό θεωρώ πως καλό είναι να έχουμε μια αναλυτική έκθεση αλλά η οποία θα είναι και αρκετά γενική. Αρκεί να αναφερθούμε μόνο σε λίγες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ε, νομίζω πως θα έχουμε και καλό αποτέλεσμα. Οι με μεμονωμένες εκθέσεις για τα μονομένα κράτη μπορούν να συζητηθούν αλλού σε, και σε άλλες συμφωνίες. Εμείς πρέπει να δούμε το σύνολο. Και αναμένω βεβαίως τις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις και θα ήθελα να πω πως θα συνεργαστούμε οπωσδήποτε και νομίζω θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόμες που εκπροσωπεί τον σκιώδη συγητή της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ε, παρακαλώ, έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε, κυρία Γκόμες. Θα μιλήσω εκ μέρους του σκιώδου συγητή μας που δεν μπορεί να είναι εδώ. Γιατί συμμετέχει σε μία αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Ταϊβάν. Πιστεύει ότι η έκθεση είναι καλή, συγχαίρει τον κύριο Μπουτικόφερ. Είναι μια ισορροπημένη βάση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε και θεωρείται σημαντικό να επικεντρωθούμε σε λίγα αλλά σημαντικά σημεία. Πιστεύει ότι θα φτάσουμε δε σε καλούς συμβασμούς. θεωρεί τα πιο σημαντικά σημεία είναι η ανανεωμένη ε, στρατηγική για την Νοτιοανατολική Ασία που αναγνωρίζει τη σχέση με την περιοχή αυτή, χρησιμοποιεί τα διάφορα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και θεωρεί ότι η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να αυξηθεί ε, στην περιοχή σε όλα τα φόρουμ και φυσικά το ΑΣΕΑΝ είναι το πιο σημαντικό από αυτά τα βήματα, από αυτά τα φόρουμ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο να αναπτύξουμε δραστηριότητες για την ανάπτυξη που συμμετέχουν όλοι, ε, τη σταθερότητα της αγοράς, ε, την κοινωνική δικαιοσύνη, ε, το διάλογο σε πολιτικούς και κοινωνικούς τομείς. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ε, να αναφερθούμε στις συμβάσεις του ILO και θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως από την, ε, τις χώρες αυτές. Επίσης, ε, οι εθνικές, οι ντόπιες εταιρείες και οι ξένες εταιρείες θα, που δραστηριοποιούνται στην ΑΖΕΑΝ θα πρέπει να σέβονται την αρχή της εταιρικής ευθύνη. Η συνεργασία με τα μέλη της ΑΖΕΑΝ πρέπει να εφαρμοστεί. Παραδείγματο χάρη για τι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κατευθυντικέ γραμμέ του ΟΗΕ είναι σημαντικό να εφαρμοστούν. Είναι σημαντικό ότι τα συνδικάτα ε, ε, εμφανίζονται σε διάφορες χώρες, παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο, περίπου στην Ινδονησία, τα συνδικάτα εργαζομένων. Σημαντικό Μέλο φυσικά λόγω του πληθυσμού τη καταρχά, λόγω των διαστάσεών τη. Αλλά υπάρχουν και άλλα μέλη τη ΑΖΕΑΝ όπου τα συνδικάτα είναι φημωμένα, δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά τον απασχολούν. Ειδικά γυναικών και κοριτσιών που είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού ε, και γενικά η ισότητα των δύο φύλων είναι μια προτεραιότητα για αυτόν. Οτιδήποτε γενικά μπορεί να προωθήσει να ανταλλαγή των φοιτητών, τι επαφέ μεταξύ των ανθρώπων και λαών, η διευκόλυνση Φερρυπίν που προφέρει το πρόγραμμα Erasmus Mundus σε οικονομικό επίπεδο, ούτω ώστε να υπάρξουν καλύτερε επαφέ μεταξύ των ακαδημαϊκών καθηγητών πανεπιστημίων της Ευρώπης και των χωρών ΑΖΕΑΝ. <coughs> Αυτά τα σημεία μου ζήτησε να παρουσιάσω, Μάικλ. Και τα οποία συμμερίζομαι και εγώ βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκόμες. Ο κύριος Βότσον τώρα στη συνέχεια. Um, uh, Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι στην ίδια κατάσταση με την κυρία Γκόμες, δεν είμαι σκιώδης ηγητής για την έκθεση, αλλά ο δικός μας ηγητής δεν μπόρεσε να είναι παρόν και επομένως τον αντικαθιστώ και εκ μέρους της ομάδας μας θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Μπουτικόφερ για μια ευρεία πλήρη έκθεση από ό,τι φαίνεται. Η ομάδα μου εντυπωσιάστηκε από μια φράση στην παράγραφο 1 όπου γίνεται λόγος για την ΑΖΕΑΝ που λέει παρά τις εσωτερικές διαφορές. Αν δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ε, θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η ΑΖΕΑΝ είχε μεγαλύτερη επιτυχία από εμά για να ξεπεράσει αυτές τις εσωτερικές τις διαφορές. Υποστηρίζουμε την πρόταση του εισηγητή να διοριστεί ένας επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΑΖΕΑΝ. Αυτό θα είναι ένα θετικό βήμα. Είναι πιο ε, είμαστε λίγο πιο σκεπτικιστές για την κοινοβουλευτική συνέλευση μεταξύ ΑΖΕΑΝ και Ευρωπαϊκή Ένωσης, γιατί από, αυτό, από την εμπειρία μας ε, με την Ανατολική Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική δεν ήταν απόλυτα επιτυχής και ευτυχής. Αλλά τέλο πάντων οποιαδήποτε επαφή μεταξύ, μεταξύ βουλευτών είναι καλύτερη παρά από τη μηδενική επαφή. Επίσης, τονίζουμε τη σημαντική τη σημασία του Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ΑΣΕΑΝ. Ε, υπάρχει εδώ και 15 χρόνια. Δεν υποστηρίζεται παρκώς από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν την ξέρουν πολύ, αλλά κάνει καλή δουλειά στην πολιτιστική ανταλλαγή, στην ανταλλαγή και επαφή των ανθρώπων, Και επειδή δεν καταλαβαίνουμε τόσο καλά του Ασιάτες όσο, όσο καταλαβαίνουμε άλλου λαού, θα θέλαμε αυτό το Ίδρυμα, το ΑΣΕΦ, να το υποστηρίξουμε όσο μπορούμε. Και επίσης καλωσορίζουμε την επιμονή του εισηγητή να υποστηρίξουμε τη δημιουργία μιας διακυβερνητικής επιτροπής για ανθρώπινα δικαιώματα στην ΑΖΕΑΝ, γιατί υπάρχουν τεράστια θέματα εδώ θέματα που αυτό το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συζητήσει α, με πολλά μέλη της ΑΖΕΑΝ. Και μπορεί να το κάνει ε, μακροπρόθεσμα πιο εύκολα από ότι με χώρες ας πούμε, της Βορειοαφρικής. Επομένως, ε, γενικά υποστηρίζουμε αυτή την έκθεση και συγχαίρουμε τον κύριο Μπουτικόφα για τη δουλειά του. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γουάσα. Ε, η κυρία Αρτίν δεν είναι. Ο κύριος Τάνοκ ε, είναι παρόν και εκπροσωπεί την ομάδα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, και οι άλλοι συνάδελφοι. Έτσι και εγώ εκπροσωπώ κάποιον, την κυρία Σουζίντε Μαρτίνη, η οποία είναι συγκήτρια των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Θα συγχαρώ και εγώ τον κύριο Μπιουτικόφερ για μια ισορροπημένη και ενδιαφέρουσα έκθεση. Μου αρέσει η γενική κατεύθυνσή τη. Προφανώς η συνεργασία με τον Αζίαν είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά για το μέλλον. 600 εκατομμύρια άνθρωποι είναι μεγαλύτερη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, είναι το μέλλον η Ασία και της οικονομίας πρέπει να έχουμε στενές σχέσεις, αλλά ο ΑΖΙΑΝ είναι και ευέλικτος οργανισμός, έχουν διάφορες συνθέσεις ε, με την Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Κίνα κτλ. και θα διευρυνθούν και προφανώς προσπαθούν να μιμηθούν έννοιες όπως η ενιαία αγορά. Τώρα δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι και το ένα νόμισμα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Μου αρέσει ιδιαίτερα η παράγραφος 14 που ενθαρρύνει την διδασκαλία των Αγγλικών. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα αγγλικά, πλέον δεν είναι θέμα των ΙΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και, και μια παραλλαγή θα έλεγα ασιατική. Και όπως ε, και ο Γκρέαμ Γουάτσον, έτσι και εγώ ανησυχώ για την παράγραφο 6, όπως άλλωστε και η Σούζη Ντεμαρτίνη, για την ιδέα μιας ε, κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Φταίω βέβαια. Πριν από μια δεκαετία στην έκθεσή μου είχα ζητήσει ε, κάτι ανάλογο με την ανατολική εταιρική σχέση, το τα λοιπά Πράγματα οποία είχαν τα καλά τους και τα κακά τους. Είναι ακριβές υποθέσεις, ε, υπερφιλόδοξες και συχνά δεν πηγαίνουν. Δεν ε, παρήσανται οι βουλευτές. Εγώ μια τέτοια νέα συνέλευση θα την δεχόμουν εάν καταργηθούν οι διμερείς αντιπροσωπείς του Κοινοβουλίου με τις αντίστοιχε χώρες. Αλλιώς θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα και θα κουράζονται και οι βουλευτές. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του μοντέλου του Κογκρέσου. Δεν υπάρχουν μόνιμες αντιπροσωπίες, αλλά μόνο ad hoc από την Επιτροπή Εξωτερικών με μέλη των άλλων επιτροπών κατά περίπτωση. Το ίδιο και για την παράγραφο 19. Τώρα αντιλαμβάνομαι πως είστε φράσινος ε, και έχετε τις ιδιαίτερες ευαισθησίες σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε πως μπαίνει στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών μελών του ΑΖΙΑΝ, ειδικά όσον αφορά το ενεργειακό και γεωργικό τους μείγμα. Νομίζω κάποιοι συνάδελφοι έχουμε συλλογογράψει με την Σούζη Μαρτίνη μια τροπολογία αλλά βεβαίω, ε, συνολικά θα υπερψηφίσουμε την έκθεση καθώ σα στο σύνολό την επιτυχία θα έλεγα. Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοφ για την παρέμβασή σας. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλα μέλη που θέλουν να παρέμβουν. Αν όχι, τότε θα ζητούσα ο εκπρόσωπο ε, τη εξωτερική υπηρεσία, ο ε, κ. Μπρίσμα να λάβει τον λόγο εξ ονόματο τη ε, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Έχετε τον λόγο κύριε Μπρίσμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Ευθυγραμμίζομαι σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι κατά την τελευταία συζήτηση. Να τονίσω ότι καλοχαιρετίζουμε την υποστήριξη για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ ΑΣΕΑΝ, στις σχέσεις αυτές που ευθυγραμμίζονται πάρα πολύ με τη δική μας προσέγγιση και καλωσορίζουμε τις προτάσεις που έγιναν για αναβάθμιση των σχέσεών μας με τις χώρες ΑΣΕΑΝ που θεωρούμε φυσικό εταίρο της ΕΕ σε αυτή την ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή περιφέρεια του κόσμου και από το 2012 υπάρχει μια πραγματική προώθηση στις σχέσεις ΑΣΕΑΝ και ΕΕ με την έγκριση ενός ε, των προγραμματών δράσης ε, και σε σχέση με την ε, συμφωνία συνεργασίας και όλα αυτά σε υψηλό επίπεδο και ανταλλαγών απόψεων και προσεγγίζουμε έτσι το να διατηρηθεί αυτή η προώθηση στην πολιτική αυτή τροχιά ώστε σε μια επόμενη υπουργική συνάντηση να διευρύνουμε τις δράσεις μας με νέους τομείς που αναφέρονται επίσης και στην έκθεση μη παραδοσιακά για παράδειγμα θέματα ασφάλειας ένα από αυτά και να δούμε και την αλληλοσύνδεση, αλληλοσυνδεσιμότητα σε σχέση με την περιφερειακή αυτή ολοκλήρωση, προσπάθεια ολοκλήρωσης σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ίσως ένα ίσονος σημασίας θέμα όσον αφορά το 25, σημείο 25. Είδαμε κάποιες τροπολογίες που κατατέθηκαν σε σχέση με την πιο ισορροπημένη διατύπωση του κειμένου και καλοδεχόμαστε αυτές τις προτάσεις. Υποστηρίζουμε πάρα πολύ αυτή την έκθεση, αυτό το έγγραφο αυτή της έκθεσης και καλωσορίζουμε τις προτάσεις. Πρόεδρε, με την έγκρισή σας να δώσω επίσης τον λόγο στον συνάδελφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρίσταται. Ευχαριστώ. Οι που προτάθηκαν στο ψήφισμα, Επιγραμμίζονται. με τη συνεργασία που υπάρχει από πλευρά Κομισιόν η Γενική μα Διεύθυνση καλωσορίζει την πρόταση αυτή, την πρόταση ψηφίσματος, ενδιαφέρουσα, ισορροπημένη Η επόμενη περίοδος ε, θα ξεκινήσει στο εγκυσμένο, το 2014. Και η κατεύθυνση που έχουμε συμφωνήσει με διάφορους ενδιαφερόμενους της ΑΖΕΑΝ ουσιαστικά πηγαίνει προς την ίδια με αυτό το κειμένο. Τρεις βασικοί τομείς υποστήριξης θα μπορούσαν να εντοπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στον ένα τομέα θα βασιστούμε στην παρελθούσα εμπειρία, περιφερειακή ολοκλήρωση και εκεί θα εφαρμόσουμε όπου μπορούμε την ευρωπαϊκή εμπειρία. Η δεύτερη συνιστόσα, η δεύτερος τομέας είναι η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των καταστροφών που αναφέρεται ρητά στο ψήφισμα. Ε, η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και με την ευαισθησία την ευπάθεια των αστικών περιοχών σε αυτήν την περιοχή του πλανήτη. Και ο τρίτος τομέας που, που προέκυψε από τις αρχικές συζητήσεις είναι ένα μέσο ε, ευραίος διαλόγου όπου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε θέματα της μη παραδοσιακής ασφάλειας, θέματα δηλαδή που ενδιαφέρουν πολύ και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και που τα ανέφερα και ο συνάδελφος από αυτήν. Ευχαριστούμε πολύ τους εκπροσώπους τη Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Επιτροπή Επιτροπής. Πρωτού δώσω τον λόγο στον συγητή κ. Μπιουτικόφερ. σω βγαίνοντα από το προσωρινό μου ρόλο του Προέδρου θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία που αναφέρθηκαν όσον αφορά την δημιουργία αυτή τη κοινοβουλευτική συνέλευση ΕΕ ΑΣΕΑΝ. Αυτό που προτείνει ο εισηγητής πιστεύω ότι είναι να αναβαθμιστεί σε πολιτικό επίπεδο η κοινοβουλευτική αυτή εκπροσώπηση, η συνέλευση. Η συνθήκη προβλέπει την δημιουργία μια τέτοιας κοινοβουλευτική συνέλευση, όπω για παράδειγμα την κοινοβουλευτική συνέλευση ΕΕΑΚΕ και για μια βάση για το Συμβούλιο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως για τη Euronest και την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Στο μέσο της εξορθολόγησης ε, των ε, κοινοβουλευτικών αυτών συνελεύσεων να είμαστε περισσότερο λειτουργικοί και λιγότερο δαπανηροί. Δεν μπορούμε όμως ε, να περιθωριοποιήσουμε μια τόσο σημαντική περιοχή του κόσμου όπως αυτή που συναποτελούν οι χώρες ΑΣΕΑΝ χωρίς το κοινοβούλιο μας όταν επικεντρώνεται στις σχέσεις με αυτές τις χώρες πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει μια κοινοβουλευτική διάσταση. Πάντα όμως μέσα σε ένα πλαίσιο που πιστεύω ότι πρέπει να είναι ορθολογικό λογικό και απλούς, α, εξαπλουστευμένο ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες. Για να απαντήσει σε ερωτήσεις που τέθηκαν, ο κύριος εισηγητής, ο κύριος Μπιουτικόφερ έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Thank again, Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, για τα σχόλια που έγιναν από κάποιους ε, συναδέλφους, ε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ε, συνεισφορά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Λάιχτφριντ βεβαίω δεν μπόρεσε να υποβάλει τροπολογίες εγκαίρως. Προσπαθώ να το διορθώσω με το να ενσωματώσω κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, αλλά θα προσπαθήσω να προτείνω και κάποιες από τις τροπολογίες του ως δικές μου για να βοηθήσω την κατάσταση. Απλά να το ξέρουν όλοι το τι θα κάνω. Κατόπιν όσον αφορά αυτό το οποίο είπε η κυρία Γέγλε για το να είμαστε γενικόλογοι. Συμφωνώ με την αρχή αυτή και εμένα αυτή ήταν η προσέγγιση μου και θα δούμε αν εφαρμόστηκε σωστά. Η προσέγγιση μου ήταν πως ε, συγκεκριμένα παραδείγματα θα αναφέραμε μόνο όπου ήταν χαρακτηριστικά και ενδεικτικά της κατάστασης. και δεν αφορούν μόνο τις ε, διμερείς ε, σχέσεις ε, μονομένων χώρων. Κατόπιν. Με προσέγγισαν διάφοροι και με ρωτούσαν γιατί αυτή η έκθεση εστιάζει τόσο λίγο στο εμπόριο. Εστιάζει τόσο λίγο στο εμπόριο, παρά το ότι είναι τόσο σημαντική διάσταση της σχέσης αυτής. Αλλά είναι αυτό το οποίο πρέπει να εξηγήσουμε όλοι σε κάθε συνομιλητή είναι πως ως ένα βαθμό δεσμευόμαστε από τις αρμοδιότητες Επιτροπής μας. Δεν είμαστε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ελπίζω να με συγχωρέσουν λοιπόν συναδελφοί για το ότι δεν ε, μίλησα πάρα πολύ ε, για το εμπόριο. Επίσης θα αναφέρω πως είχα την ευκαιρία στο τελευταίο Στρασβούργο να συναντηθώ και με τους 10 πρέσβεις του Αζίαν και να μιλήσουμε για το σχέδιο έκθεσης και θα πάρα πολύ καλές αντιδράσεις και σχόλια και κάποια από αυτά βέβαια θα εξετάσουμε σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τάνοκ στις γενικές γραμμές θα συμφωνούσα μαζί σας για τις αντιπροσωπείες και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να καταργήσουμε τις αντιπροσωπίες, όμως ε, αν θα το ήθελαν οι υπόλοιποι αλλά στη σύγκριση που έγινε με άλλες περιοχές θα έπρεπε να είμαστε κάπως ευαίσθητοι όσον αφορά το διπλωματικό πλαίσιο αν έχουμε διακοινοβουλευτικές διασκέψεις με διάφορες περιοχές και θέλουμε να πούμε πως παίρνουμε στα σοβαρά την περιοχή του Ατζίαν. Δεν πρέπει να στείλουμε κανένα μήνυμα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Με το να μην έχουμε μεικτή κοινοβουλευτική διάσκεψη. Οπότε επίσης κάπου θα συμφωνήσουμε. Τέλος, όσον αφορά τη διάσημη διαβόητη παράγραφο 25 σας υπόσχομαι πως ε, θα προσφέρω, θα υποβάλω διαφορετικές διατυπώσεις και ελπίζω να ικανοποιηθούν όλοι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπιουτικόφερ. Σημειώσαμε τις παρατηρήσεις των συναδέρφων. Και δεν ξέρω κύριε Σίγητα αν δεδομένου των ανταλλαγών απόψεων που είχαμε, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε, κύριε Κόφερ την ημερομηνία της ε, δεύτερης συνόδου του Οκτωβρίου για να ψηφιστεί η έκθεση στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε αυτό, κύριε Σιγητά, τι λέτε. Στην Σύνοδο Οκτωβρίου 2 ψήφιση, έγκριση, προς έγκριση. Πολύ καλά. Αν συμφωνείτε περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης που είναι η συμφωνία ε, σύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας. Ξέρετε το 2004 το Συμβούλιο Υπουργών έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαπραγμάτευση μιας τέτοιας συμφωνίας με την Ινδονησία. Ολοκληρώθηκαν το 2007 αυτές οι διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία υπεγράφει το 2009 και τώρα το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στην έγκριση αυτής της συμφωνίας. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ κάτι. Τη μεγάλη διαρροή χρόνου που πέρασε μεγάλο χρόνο που πέρασε από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες για αυτή τη συμφωνία και από την, μέχρι την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτών. Ε, είναι πολύ μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το συντμίσουμε, να το συντομεύσουμε γιατί υπονομεύουν την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιες καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να τονίσω τη σπουδαιότητα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Δημοκρατία της Ινδονησίας με πάνω από 200 εκατομμύρια ε, κατοίκων με το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό και γι' αυτό αυτή η συμφωνία έχει τεράστια σπουδαιότητα. Και όπως και σε άλλες τέτοιες συμφωνίες σύνδεσης, παρακολουθήσαμε ακολουθήσαμε το πρότυπο μιας προσωρινής έκθεσης interim report όπου θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα θέματα, τα ενδεχόμενα προβλήματα τα οποία μπορεί να τίθενται για μια τέτοια συμφωνία και τις προτεραιότητες. Ανοίγουμε μέσω στη συζήτηση και δίνω τον λόγο γι' αυτό στην εισηγήτρια τη συνάδελφο Ανά Γκόμες για να μας παρουσιάσει ακριβώς την έκθεσή της. Παρακαλώ κυρία Γκόμες, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η διαφορά που τονίσατε ανάμεσα στην υπογραφή της ε, συμφωνίας μέχρι την τελική επικύρωση από το Κοινοβούλιο και την εφαρμογή της οφείλεται στην ε, διαδικασία επικύρωσης. Μου είπαν ότι 26 από τα όχι, διαφωνεί η μιλήτρια. 25 από τα 28 κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι δύο κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει. Η Κροατία είναι στη διαδικασία επικύρωσης. Ελπίζω να μου απαντήσει, να μου πει κάτι σχετικό η Κομισιόν ή το Συμβούλιο για το ποια είναι η δυσκολία την οποία προσκρούν οι εθνικέ διαδικασίες επικύρωσης, γιατί πραγματικά είναι αργή αυτή η διαδικασία. Και είναι αργή γιατί η Ινδονησία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλα τα συμπαρουμαρτούντα. τακτικέ επισκέψεις. Είναι κρίμα που ο πρόεδρο τη ε, Κομισιόν και είπατε εκπρόσωπο, ε, που ε, υποθέτω επισκεπτόντουσαν την Ινδονησία δεν το έκαναν. Είναι μια χώρα που είναι ιδρυτικό μέλο τη ΑΖΕΑΝ, μόλις συζητήσαμε την ΑΖΕΑΝ. Τι θα ήταν η ΑΖΕΑΝ χωρίς την Ινδονησία. Είναι μέλο του IOC, του G20 και μια πολύ σημαντική χώρα από πολλές απόψεις. Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Ινδονησία είναι εικόνα των προβλημάτων που προκάλεσε το τσουνάμι και που οδήγησε σε ανθρωπιστική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνης περιοχής. Επίσης το πρόβλημα ε, της σύγκρουσης στο ΆΤΣΕ, εσωτερικό πρόβλημα της Ινδονησίας. Στέλνουμε εκλογικές αντιπροσωπείες στην Ινδονησία εδώ και χρόνια, ε, οι οποίες αξιολογούν, δηλαδή παρατηρητές ε, στι εκλογές, που αξιολογούν τη διαδικασία των εκλογών και οι δίκαιες ε, και ανώθευτες εκλογές ε, είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Είναι μια νεαρή δημοκρατία που έζησε πολλά χρόνια έζησε πολλά χρόνια κάτω από στρατιωτικό ζυγό και το 1989 έγινε δημοκρατία. Και είναι εντυπωσιακή η πρόοδος που έγινε αυτό το μεσοδιάστημα από τους Ινδονήσιους στον τομέα της δημοκρατίας. Είναι σημαντική αυτή η χώρα για την δημοκρατία και είναι η χώρα με το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Και είναι η απόδειξη ότι η δημοκρατία και το Ισλάμ είναι απόλυτα συμβατά. Πολλοί το αρνούνται, αλλά να που το παράδειγμα της Ινδονησίας το διαψεύδει. Αυτή η συμφωνία, η, ειρηνευτική συμφωνία και η συμφωνία συνεργασίας είναι πολύ ευρεία, πολύ σημαντική. Θέλει να ενταθούν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ανωσυνδονησίας, όχι μόνο οικονομικές, που ούτως ή άλλως αναπτύσσονται γοργά. Τα τελευταία έξι χρόνια οι εξαγωγές μας προς την Ινδονησία διπλασιάστηκαν. Είναι μια χώρα με πολύ νεαρό πληθυσμό και με μια μεσαία τάξη που αυξάνεται, που έχει τρομερό δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης οι επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδονησία ανθούν και οι Ινδονήσοι παραγγέλνουν πολλά αεροπλάνα και, άλλα, και άλλους εξοπλισμούς από τους Ευρωπαίους. Επομένως, πραγματικά στον οικονομικό τομέα οι σχέσεις αναπτύσσονται, αλλά θα πρέπει οι σχέσεις αυτές να συνοδευτούν από ανάπτυξη και των πολιτικών σχέσεων. Καλό είναι που αυτή η συμφωνία έχει ε, βασικό στοιχείο τα άρθρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την, κατα... την καταπολέμηση των όπλων μαζικής καταστροφής, επίσης ε, να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα των χωρητών όπλων και του λαφρύ οπλισμού, όλα αυτά που βρίσκονται στην χάρτα του ΟΗΕ Αυτά αναφέρονται και στην ε, νέα συμφωνία. Φυσικά είναι νεαρή δημοκρατία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα στην Τονισία και στην Ευρώπη. Υπάρχουν και ή προβλήματα, παρότι μερικέ από τι δημοκρατίε μα είναι από τι πιο παλιέ στον κόσμο. Και πολλά μπορούμε να κερδίσουμε αν έχουμε πιο έντονες σχέσεις. Η Ινδονησία παίζει ρόλο, όπως αναφέρθηκε, σημαντικό στην ΑΖΕΑΝ, ε, εξαπλώνοντας τις ε, τις δημοκρατικές αρχές. Παραδείγματο χάρη, δέστε ε, τη Μιαμάρ που εξελίσσεται και που στρέφεται προς την Ινδονησία ε, ως πρότυπο, για να τη δει πρότυπο. Πραγματικά μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο του προτύπου στις άλλες χώρες της περιοχής. Είναι σημαντικός εταίρος για τους παγκόσμιου παγκόσμιους προβληματισμούς για την ασφάλεια και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας αλλά και παγκόσμια. Και ένας άλλος τομέας είναι η ασφάλεια τη θάλασσες. Αλλά όλα τα προβλήματα για με το ξύλο, την κλιματική αλλαγή κτλ. είναι σημαντικός ο ρόλος της. Φυσικά υπάρχουν τομείς προβληματικοί γιατί πολλές τάσεις στον κόσμο και στο μουσουλμανικό κόσμο ειδικά. Φυσικά υπάρχουν και στην Ινδονησία, ε, υπάρχουν κάποιες ε, εξτρεμιστικές ομάδες και εκεί. Υπάρχουν προβλήματα στην Ινδονησία λοιπόν. Το να συνεργαστούμε με την Ινδονησία για την καταπολέμηση της δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα θυμάστε τον βομβαρδισμό στο Πάλι και άλλες βόμβες που έσκασαν στην Ινδονησία και τότε συνεργάστηκαν οι Ινδονήσοι με, ξένους, με τους ξένους. Επίσης, μην ξεχνάμε το πρόβλημα της ανάκτησης κλεμμένων προσόδων, ε, καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχει ένα πρόβλημα αυτό στη χώρα. Ε, και αυτό συνδέεται και με την διακυβέρνηση των ε, εταιριών. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ πήγα πρόσφατα στην Ινδονησία και ήμουνα πρέσβης στην Ινδονησία όταν ε, άνοιξε στη δημοκρατία, τα πρώτα χρόνια που έγινε δημοκρατία ε, η Ινδονησία. Και οι ακτιβιστές και οι οργανώσεις της, για τα ανθρώπινα δικαιώματα θυμάμαι πώς ήταν και πώς είναι τώρα, πώς αναπτύχθηκαν. Υπάρχει ελευθερία του τύπου, υπάρχει ζωτικότητα, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε με τη χώρα αυτή. Και χαίρομαι που τα μέλη του Ινδονησιακού Κοινοβουλίου, όταν άκουσαν ότι εμείς θέλουμε να γράψουμε αυτή την έκθεση, προσφέρθηκαν να έρθουν εδώ και να συζητήσουν μαζί, μαζί μας για όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν και που αναφέρουμε στην έκθεση. και θέλουν αυτή η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία να χρησιμοποιηθεί για να προωθηθούν οι σχέσει. Τα πιο περίπλοκα θέματα είναι τη διαφθορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, βεβαίω. Είδαμε τις ε, τρομοκρατικές απόπειρες είναι μια πολύ όμορφη κοινωνία και χώρα. Εθνικά, γλωσσικά, θρησκευτικά. Αλλά επειδή δεν είναι απομονωμένο κάστρο αυτή η χώρα, και ειδικά επηρεάζεται από τα τεκτενόμενα στο μουσουλμανικό κόσμο, έχουμε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, βεβήλωση των εκκλησιών, υπάρχει το πρόβλημα της παππούα που συνεχίζεται και όπου χρειάζεται πιο έντονος διάλογος. Και οι συνάδελφοί μας από την Ιδονησία είναι διατεθειμένοι να τα συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα. Κάτι που είναι θετικό βέβαια. Τελειώνοντας, να τονίσω ότι αυτή η συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασίας θα συμπληρωθεί από μια συμφωνία οικονομικής συνεργασίας οικονομική εταιρική σχέση, συγγνώμη, η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή και που σκοπό έχει να άρει διάφορα εμπόδια που υπάρχουν ε, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στις προμήθειες. Και πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασία θα εντείνει τις σχέσεις μας με την Ινδονησία και όλοι θα κερδίσουμε από αυτό. Είναι μια στρατηγική σημασία χώρα και πρέπει να είναι εταίρος μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Συγγήτρια. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας τον λόγο στους κοιόδης εισηγητές των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Ομεν Ρόιτεν πρώτη. Έχετε τον λόγο. Ehm, ναι. Θα ξεκινήσω με τις ευχαριστίες προς την κυρία Γκόμες και για αυτά τα οποία μας είπατε. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η πρώτη ε, συμφωνία με μια χώρα του Αζίαν και αυτό οφείλεται στο ότι όχι μόνο είναι μια φανταστική χώρα η Ινδονησία αλλά ε, και δυναμική και το είπε αυτό η Άννα και πράγματι θέλουμε να έχουμε καλές ε, διμερείς σχέσεις με την μεγάλη αυτή χώρα και πρέπει να έχουμε. Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία αφορά α, ε, τις ε, οικονομικές, πολιτικές και τομεκές ε, εξελίξεις και θέλουμε βέβαια να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα και το είναι σωστό γιατί είναι μια κατάσταση αμοιβαία υποφελής και έτσι πρέπει να είναι και Ινδονησία και για εμάς. Είναι καλό και για τους Ινδονήσιους αλλά και για τους Ευρωπαίους. Και θεωρώ πως στην έκθεση που παρουσίασε η Άννα, σύμφωνα νομίζω υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να εμφανιστούν καλύτερα η διαφθορά, σεβασμός θρησκευτικών μειονοτήτων, η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών. Ε, είναι καλό βεβαίως το να τα προσέχουμε αυτά γιατί βεβαίως μια τέτοια συμφωνία βασίζεται και σε αρχές που έχουμε. Ισότητα, αμοιβαίως σεβασμός, δημοκρατία, κράτος δικαίου δικαιώματα ατομικά και συλλογικά και είπα και με τον το είπα στον πρέσβη την προηγούμενη εβδομάδα πως πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα να κοιταχτείτε στον καθρέφτη για να δείτε πως μπορεί να απτυχθεί περαιτέρω η χώρα αλλά κατόπιν αν δούμε πως ο καθρέφτης είναι καλός, θεωρώ πως η έκθεση σε κάποια σημεία δεν λαμβάνει υπόψη τις ε, πλανθασμένες εξελίξεις που ε, είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν ελλείψεις, αλλά πώς μπορούμε να δούμε και τα θετικά. Να τα τονίσουμε περισσότερο όχι μόνο για να ικανοποιήσουμε τους ανθρώπους, αλλά να μην περιγράφουμε και τα αρνητικά μόνο. Γιατί να δώσουμε και την αίσθηση ότι υπάρχει μια πρόκληση για βελτίωση. Και θα συνεργαστούμε τώρα με την Άννα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Να είναι επικοδομητική η έκθεση, ισορροπημένη, αλλά πρέπει βεβαίω να υπάρξει, όπως είπα, και αυτός ο χαρακτήρας της πρόκλησης για να επιτύχουν το κάτι καλύτερο. Και βεβαίω αυτό νομίζω πως θα μας οδηγήσει τελικά σε μια καλή ε, συμφωνία. Και αναμένω πράγματι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών κύρωσης στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Ε, ε. Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Ομερόιτεν. Τώρα ο κύριος Βότσον παρακαλώ. Thank you, Chairman. I too... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Άμα την Άννα Γκόμες για την έκθεσή της και συμφωνώ με αυτά που είπατε στην αρχή. Το 2007 μονογράφηκε η συμφωνία, ε, υπογράφηκε το 9 και ακόμα είναι μπροστά μας. Έχει κρατήσει πάρα πολύ διαδικασία. Χρειαζόμαστε ε, δράση στο Συμβούλιο. Να πιέσουμε τις χώρες στο Συμβούλιο που δεν το έχουν κάνει να το κάνουν. Ούτε η Γαλλία ούτε η Ελλάδα έχουν ε, επικυρώσει τη συμφωνία. Φυσικά και η Κροατία μέσω παραρτήματο θα πρέπει να, το, να την επικυρώσει. Σε μια τέτοια εποχή υψηλή ανεργία στην Ευρώπη, ε, είναι απαράδεκτο να καθυστερούμε την υπογραφή μια τέτοια συμφωνία που θα είναι υποφελή και για όλα τα κρατη και θα φέρει δουλειέ και επενδύσει. Ε, θα κερδίσουμε πάρα πολλά από αυτή τη συμφωνία και θα πρέπει οπωσδήποτε να ανασκομποθούμε για να αποφύγουμε τέτοιες καθυστερήσει. Ένα από τα πράγματα που αρέσει στην ομάδα μου στην έκθεση είναι ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδονησία. Ήταν ε, επιτυχή ε, πρωτοβουλία. Τρίτη φορά γίνεται με τους Ινδούς. Για δεύτερη φορά ε, έχουμε καθυστερήσει τις ε, συζητήσεις, οι Ινδοί δηλαδή, με δική τους πρωτοβουλία καθυστέρησαν τις συζητήσεις και η στάση της Ινδονησίας δείχνει ότι ενδιαφέρεται να βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη τη χώρα. Συμφωνώ με την Αναγκόμες ότι ο πρόσφατος νόμος για τις ε, οργανώσεις, μαζικές οργανώσεις θα μπορούσε να είναι πρόβλημα για την κοινωνία των πολιτών μακροπρόθεσμα και τις οργανώσεις της. Αλλά θα πρέπει να δούμε την επίπτωση αυτού του νόμου. Υιοθετήθηκε πριν από λίγους μήνες και είναι ασαφές ακόμα πώς θα επηρέασει τα πράγματα και θα προτιμούσαμε βέβαια να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να δούμε τι θα συμβεί. Συμφωνούμε επίσης με την ανησυχία της Άννας για τις θρησκευτικές νότες, Μιλάμε για μια χώρα όπου η θρησκευτική ελευθερία εξασφαλίζεται από το Σύνταγμα, αλλά και η κυβέρνηση Ινδονησία θα αναγνώρισε ότι χρειάζεται και άλλε προσπάθειε για να προωθηθεί η ανεξιθρησκεία. Και δεν μιλάω μόνο για τους χριστιανούς, ε, ούτε για τους οπαδούς τη Αχμαντίγια, Συχνά δεν υπάρχουν προβλήματα σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά η πραγματικότητα σε τοπικό επίπεδο, όπως εφαρμόζονται οι πολιτικέ, εκεί είναι το πρόβλημα. Αναγνωρίζουμε ότι έχει συνήθει πρόοδο, βέβαια, παρά το γεγονό ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, η κυβέρνηση ασχολείται. Φυσικά ανησυχούμε στην ομάδα μου, όπως και άλλες ομάδες, ε, με το φαινόμενο, για το φαινόμενο της διαφθοράς και το ξέπλυμα του χρήματος σοβαρό θέμα είναι αυτό, όπως και ο συνεχιζόμενος ρόλος και η εμπλοκή των, ε, του στρατού στην οικονομία, των ενόπλων δυνάμεων στην οικονομία. Αλλά δεσμεύτηκε η Ινδονησία στο G20 να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα με αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους φόρους φορολογική διαφάνεια δηλαδή. Θα πρέπει να αναγνώσουμε αυτή την πρόοδο. Επίσης, ε, οι πρόσωποι των ε, εγκληματικών οργανώσεων καταλήγουν καμιά φορά εξάγονται από τις οργανώσεις αυτές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω σε αυτές τις συζητήσεις με την Ινδονησία να υπάρξει πρόοδο και για αυτό το θέμα. Υπάρχουν τρεις μικροί τομείς όπου θα θέλαμε να πούμε περισσότερα στην έκθεση και θα κάνω προτάσεις για αυτούς. Ο ένα είναι να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο εμπόριο και επενδύσει. επενδύσεις. Δεύτερος τομέας να δώσουμε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της ενέργεια και ιδίως στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι έχει μαζικό δυναμικό που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα και να αναπτύξουμε συνεργασία στον τουρισμό και στις μεταφορές καθώς ε, και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά εκεί για να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές για την διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι νοικιό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούν για την καταστροφή των κοραλιών ε, με τη χρήση δυναμίτη από ψαράδες, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς που μπορούμε να εξετάσουμε ε, και όλοι μπορούμε να υποφεληθούμε από επίσημη ανταλλαγή αξιωματούχων, ας πούμε, αλλά και από ανταλλαγή απλών ανθρώπων. Θα πρέπει αυτή η ανταλλαγή δεύτερη να ενταθεί. Μην ξεχνάμε εδώ τη σημασία του, των υποτροφιών του Εράσμος Μούντους, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουμε περισσότερο την ανταλλαγή αυτή που είναι τόσο... Και αυτές οι ανταλλαγές μια τόσο γοητευτική και πλούσια με όλους τους όρους χώρα είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε κύριε Βότσον. Ο κύριος Μπιουτικόφερ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου σε όσους συνεχάρισαν την αναγκόμεση για αυτό το σχέδιο εκθεσής. Πορευόμαστε σε παρόμοια κατεύθυνση σε μεγάλο βαθμό. Όπως είπαν εκτενέστερα οι συνάδελφοι και τοποθετήθηκαν εκτενέστερα, εγώ μπορώ να είμαι συντομότερος. Να φέρω τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, είμαι βέβαιος ότι η κύρια επικέντρωση αυτής της έκθεσης είναι να <clears throat> προαχθεί η εταιρική σχέση και να μπορέσει αυτή να αναπτυχθεί μεταξύ ΕΕ και Δονησίας Δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα θεωρηθούμε υπερβολικά και δαιμονευτική απέναντι στους Ινδονήσιους. Και πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε μήπως μπορούμε να βρούμε ίσως και μια κάποια κοινή βάση ως θεμέλια για την ένταξη της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιουτικόφερ. Θα ήθελα να ξέρω, υπάρχουν άλλα μέλη που θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Άννα που γνωρίζει σαφώς πολύ καλά αυτή τη χώρα την Ινδονησία. Όταν ξεκίνησε ήταν επικεφαλής των Πορτογάλων όσον αφορά τα συμφέροντά τους και όσον αφορά και την πρεσβεία και το θέμα στην, του Ανατολικού Τιμόρ όλα αυτά πολλά λέγουν για την οριμότητα της Ινδονησίας που στο τέλος τέλος ε, εγκατέλειψε ε, την αμφισβήτηση του Ανατολικού Τιμόρ και δέχθηκε την ε, νομιμότητα αυτού του νέου κράτους. Μακάρι να μπορούσαν και άλλες χώρες να ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία. Η έκθεση είναι πραγματικά πολύ ισορροπημένη και για την Ινδονησία που είναι μια τόσο τεράστια χώρα και όσον αφορά και τον πληθυσμό της και την οικονομική της ανάπτυξη δεν μπορεί να αγνοήσει με κανένα τρόπο λοιπόν η ε, ΕΕ την ανάπτυξη των σχέσεων και καλλιέργεια των σχέσεων με την Ινδονησία σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στους τομείς ε, των οικονομικών σχέσεων και τα θέματα της δημοκρατίας επίσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την δημιουργία ε, δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ μας. Ε, είναι σημαντικό αυτό. Υπήρξαν προβλήματα σε σχέση με την Ινδονησία όσον αφορά μειονοτικά ζητήματα. Είχαμε και ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου όσον αφορά ε, την κοινότητα των μουσουλμάνων ε, Αχμαντί και σε σχέση με τις τη βελτίωση των, ε, την, της κατάστασης και σε σχέση και με τους εκπροσώπους αυτής της κοινότητας στο Λονδίνο. Αυτά τα οποία όμως παρακολουθούν και ακολουθούν οι Ινδονήσοι και με την κυβέρνησή τους επειδή υπάρχει μια παράδοση ιστορικά μιας πιο μετριοπαθούς ε, σουφιστικής παράδοσης ε, και την αντιμετώπιση των ακραίων και τζιχαντιστών που χρησιμοποιούν και τους ε, ε, ουλεμά, τους ε, ε, θρησκευτικούς δασκάλους σε σχέση με μηνύματα τα οποία αποστέλλονται για το ότι οι θέσεις αυτές είναι ασύμβατες με την παραδοσιακή μουσουλμανική, το παραδοσιακό μουσουλμανικό δόγμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενθαρρύνουμε και όλα αυτά νομίζω συνοψίζουν ότι είναι μια πολύ ισορροπημένη έκθεση για μια πάρα πολύ σημαντική χώρα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Ιδονησία θα ήθελα κάποτε να πάω εκεί. Η σχέση μας είναι πάρα πολύ σημαντική σημαντικές λοιπόν και υποστηρίζουμε <clears throat> την ανάπτυξη των σχέσεων και την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Αν δεν υπάρχουν άλλα μέλη που να θέλουν να παρέμουν και προτού δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Σούνε της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να μας δώσει κάποια δήλωση ή τοποθέτηση Προτού λοιπόν δώσω τον λόγο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, προτού πάτε τον λόγο, θα ήθελα να με παρακολουθήσετε, θα ήθελα να διατυπώσω μια ερώτηση στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα που μας διαβίβασε η συγγήτρια, που μας πρότεινε η συγγήτρια και το γεγονός ότι ήδη 25 κοινοβούλια των κρατών μελών έχουν προχωρήσει στην επικύρωση της συμφωνίας, θα ήθελα να γνωρίζω ποιοι είναι οι λόγοι ουσιαστικά για τους οποίους καθυστερήσαμε τόσο πολύ στο να προχωρήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση αυτή η συμφωνία. Έχουμε και ένα εμπορικό τμήμα αυτής της ε, πτυχής και πέρα από τις διαρκείς εκκλήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προηγούμενα να μπορεί να γνωμοδοτήσει είχαμε την ίδια εμπειρία και με άλλες συμφωνίες σύνδεσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εγκρίθηκαν πέρυσι το Δεκέμβριο συγκεκριμένα με την Συμφωνία Σύνδεσης με την Λατινική Αμερική και σε σχέση με τη Συμφωνία με την Κολομβία που το 2010 ολοκληρώθηκαν και μόνο κατά τα τέλη του 2012 μπόρεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί και να, εγκρίνει. Θα ήταν ευκταίο αυτές οι συμφωνίες όταν πραγματικά θα ολοκληρώνονται και θα πρέπει να επικυρωθούν να μπορούν να υποβάλλονται άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να μπορεί να δώσει την σύμφωνη γνώμη του, τη συμφωνία του. Ο κύριος Σουνές έχει τον λόγο παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στην τελευταία ερώτηση πρώτα. Δεν μπορώ βεβαίω να εκπροσωπήσω εγώ τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς έχει καθυστερήσει η διαδικασία κύρωσης συμφωνίας, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω είναι πως η Κροατία δεν χρειάζεται να κυρώσει τη συμφωνία. Γιατί νομίζω πως ε, υπάρχει μια παρεξήγηση ότι χρειάζεται η Κροατία να κυρώσει συμφωνία. Δεν, δεν χρειάζεται. Επίσης, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και να σας συγχαρώ για το ότι ε, τόσο γρήγορα αντιμετώπισε το ζήτημα της Ινδονησίας. Νομίζω πως ε, και το Συμβούλιο το ίδιο έκανε και είναι μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στην Ινδονησία και αυτό φάνηκε και στη συζήτησή σας. Σημαντικό είναι λοιπόν πως είναι μια χώρα κλειδί η Ινδονησία σε μια περιοχή κλειδί και νομίζω πως αναγνωρίζουμε πως ο Αζίαν χωρίς την Ινδονησία δεν θα ήταν ο ίδιος οργανισμός. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω πως η συμφωνία αυτή αν και όταν κυρωθεί θα είναι η πρώτη συμφωνία αυτού του είδου μετά τη Λισαβόνα. Ήταν και η πρώτη επίσης που είχε υπογραφεί με την Νοτιοανατολική Ασία, ε, προκαιρού βεβαίως. Θεωρώ λοιπόν πως ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, θεωρεί την Ινδονησία μια πάρα πολύ σημαντική χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδονησία έχουν πολλές κοινέ αξίες και ιδανικά και έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο σχέσεων. Και αυτό νομίζω φαίνεται στην έκθεση της κυρίας Γκόμες, η οποία είναι μια ισορροπημένη έκθεση και συμφωνούμε πλήρως με πολλά στοιχεία της. Επίσης, σημαντικό είναι να τονίσουμε πως η συμφωνία θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε το περιθώριο τομεακής συνεργασίας. Άκουσα κάποια πράγματα όπως η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή. Παράδειγμα χάρη για την κλιματική αλλαγή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδονησία είναι νομίζω προοδευτικές χώρες στο θέμα αυτό. Η συμφωνία αυτή λοιπόν μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας. Ένας άλλος τομέας που γνωρίζω καλύτερα είναι ο τομέας της εξωτερικής πολιτικής. Μπορούμε να συζητήσουμε ζητήματα όπως η Μιαμάρ, οι Ροχίνγκια οι οποίοι πηγαίνουν στην Ινδονησία από την Βυρμανία. Η Αραβική Άνοιξη καθώς ε, η Ινδονησία ήταν μία από τις ε, πρώτες χώρες που προσεκλήθησε στο Κάιρο. Με τη συμφωνία αυτή λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι πως δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Οι συμφωνίες αυτές είναι ένα πλαίσιο αναφοράς και σημασία έχει το περιεχόμενο του διαλόγου και δεν σταματάει εδώ πέρα η υπόθεση αυτή. Όλοι και το Κοινοβούλιο, οι συνάδελφοί μου στην Κομισιόν, ειδικά σε κάποια τομιακά ζητήματα, όπως τον τουρισμό, την ναυτική συνεργασία. Οι συνάδελφοι λοιπόν θα μπορεί να εργαστούν επί του θέματος. Επίσης θέλω να τονίσω πως όσον αφορά την διαδικασία ακύρωσης, γεγονός είναι πως δύο κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα ακυρώσει τη συμφωνία, αλλά ε, σας διαβεβαιώ πως ε, δεν σημαίνει τίποτα για την Ινδονησία αυτό. Ε, από ό,τι μας είπαν είναι ζητήματα εσωτερικών διαδικασιών. Οπότε δεν πρέπει να αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Τέλος, θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά το ότι αναμένουμε την ε, κύρωση της συμφωνίας και βέβαια η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου παίζει εδώ πέρα ένα ρόλο κλειδί και αναγνωρίζουμε το πόσο καλά χειρίστηκε το Κοινοβούλιο το θέμα αυτό και να συγχωρούμε την Αναγκόμες για την ισορροπημένη της έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις πολύ επικοδομητικές παρατηρήσεις τους και προσέγγιση τους για αυτή την έκθεση. Και προφανώς όπως γνωρίζετε υπάρχουν κάποια όρια σε σχέση με θέματα που μπορούν να διατυπωθούν. Έπρεπε να αφαιρέσω το δυνατόν περισσότερα και γι' αυτό έχει αυτή τη μορφή αυτή η έκθεση. Και γι' αυτό είναι, ίσως μη δεν είναι τόσο ισορροπημένη όσο θα ήθελα εγώ σε σχέση με, τις, με τα θέματα της ε, κυρίας Όμερ Ρόιτεν για παράδειγμα. Θα ήθελα να είμαστε πιο επικοδομητικοί. Και με τις τροπολογίες και συνεργασία των συναδέλφων σίγουρα θα μπορέσουμε να, να δημιουργήσουμε σωστή, το σωστό ύφος και την σωστή διατύπωση επισημένοντας το μίσο που πραγματικά η συνεργασία θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη. Όχι μόνο σε έναν από τους εταίρους αλλά και στους δύο αμφότερους εταίρους. Πράγματι δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι και οι δύο θα ωφεληθούμε και η ΕΕ και η Ινδονησία από αυτούς τους τομείς ακόμα και από τους πιο ακαθόδεις και περίπλοκους ε, τομείς που πρέπει να ε, μπορέσουν να ε, λάβουν σάρκα και οστά και να υλοποιηθούν. κατά τη της διαφθοράς, πολέμηση των φορολογικών παραδείσων, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας αυτή τη στιγμή. Και ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να συναγάγουμε από τη σημερινή κρίση. Υπάρχουν τομείς που μπορούμε να μάθουμε από τους Ινδονήσιους. Η Ινδονησία είναι μία από τις χώρες που έχει επικυρώσει την σύμβαση όσον αφορά τους μετανάστες και τι τις οικογένειές τους και την προστασία μεταναστών και οικογενειών του και πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Τα, η Ινδονησία είναι μια πραγματιστική ρεαλιστική χώρα όσον αφορά την προσέγγιση των θεμάτων των προσφύγων και συνεργάζεται πολύ καλά με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Θα μπορούσα να φανταστώ λοιπόν ότι κατά το μελλοντικό διάστημα με την επόμενη κυβέρνηση στην ε, Αυστραλία ίσως θα έπρεπε αυτές τις δυσκολίες να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, να βοηθηθεί η ε, Ινδονησία σε αυτά τα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να μάθουμε από αυτές τις ε, διεργασίες και όπως αναφέρθηκε και στους τομείς, για παράδειγμα, των κλιματικών αλλαγών και για τα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των ανανεώσιμων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας. Πέρα από άλλους τομείς και τομεακές πολιτικές που <clears throat> σωστά αναφέρονται και στην έκθεση της ε, Κομισιόν συμπεριλαμβάνονται. Είναι εκπληκτική η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από την Ινδονησία στην καταπολέμηση της πειρατείας κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με συνεργασία με τις άλλες χώρες της περιφέρειας. Και θυμάμαι όταν ήμουν εκεί κατά την αρχή της ε, δεκαετίας του 2000 ήταν ένα σοβαρότατο πρόβλημα η πειρατεία. Τώρα έχει αντιμετωπιστεί, έχει διευθετηθεί χάρη στην πραγματιστική και ρεαλιστική αποτελεσματική προσέγγιση. Πολλά μπορούμε να συναγάγουμε και να μάθουμε από πλευράς μας σε σχέση με τη, τους Ινδονήσιους και τη συνεργασία με τους Ινδονήσιους για αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και κάποιες διορθωτικές προτάσεις και εγώ ίδια θα καταθέσω τροπολογίες στην έκθεσή μου. Πολλά πράγματα που έπρεπε να αφαιθούν εκτός έκθεσης, πρέπει να παραμείνουν εκτός έκθεσης λόγω περιορισμών όσον αφορά την έκταση της ε, έκθεσης αυτής, αλλά και διορθωτικά όσον αφορά τον διάλογο για διάφορα θέματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδονησίας ακόμα και πριν αρχίσει να ισχύει η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Και εν κατακλείδη σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχει ένας τομέας που πρέπει να διευρυνθεί περισσότερο σε αυτήν την έκθεση. Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η Ινδονησία στην ευρύτερη περιοχή και για το Φόρουμ Δημοκρατίας του Μπαλί που ξεκίνησε με τις δράσεις της ε, ε, Ινδονησίας με μια ημερήσια διάταξη για τα θέματα δημοκρατίας πάρα πολύ σημαντική και όσον αφορά και τα όσα συμβαίνουν και στη Βυρμανία, Μιανμάρ αλλά και σε σχέση με άλλους τομείς ε, η Ινδονησία είναι πάρα πολύ σημαντική και πολλά μπορούμε να επωφεληθούμε από τη συνεργασία με την Ινδονησία και συμφωνώ τα μέγιστα με αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Μπιουτικόφερ ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε τη σωστή διάσταση όπως απαιτείται στην κοινωνία των πολιτών εντάσσοντας αυτή τη συνιστόσα στην έκθεση και σε σχέση και με την ε, ε, αποδοχή του κράτους ε, δικαίου και ένομης τάξης και βλέποντας ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι φόβοι ή ε, ποια προσέγγιση ακολουθείτε πρέπει να βρούμε μια επικοδομητική διατύπωση. Είναι ένα μέλημα, μια ανησυχία που υπάρχει σε σχέση με την Ινδονησία από σημαντικούς τομείς της κοινωνίας των πολιτών. Και σίγουρα θα μπορούσαμε να βρούμε ένα επαρκές πλαίσιο, ένα ενδεδειγμένο πλαίσιο για να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτή την πτυχή με το σωστότερο αποτέλεσμα. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω σε αυτή τη φάση. Εκτιμούμε την υποστήριξη που μας δόθηκε από όλους τους συναδέλφους και προσβλέπουμε στο να δούμε τις τροπολογίες τους. Και επίσης ε, με την ε, αμφίδρομη σχέση και δράση με τους ε, Ινδονήσιους συναδέλφους που θα προσέλθουν και να έχουν επαφές μαζί μας. Ο Ινδονήσιος πρέσβης, για παράδειγμα, με τον Ινδονήσιο πρέσβη που ε, έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Προσβλέπουμε λοιπόν στα σχόλια αυτά και παρατηρήσεις ε, και τροπολογίες ώστε να μπορέσει να δώσει ερεθίσματα η έκθεση ώστε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμα να μπορέσουν το γοργότερο να επικυρώσουν και να αρχίσει να ισχύει αυτή η συμφωνία το δυνατόν γοργότερα. Είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό για τη σχέση μας με την Ινδονησία. Ευχαριστούμε. Άννα. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον πρέσβη της Ινδονησίας που παρακολουθεί τις εργασίες μας. Υπενθυμίζω προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 10 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι κατάθεση τροπολογιών. Περνάμε αν συμφωνείτε στο 6 της ημερησίας διάταξής μας που είναι η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Αρμενίας για τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αρμενίας στα προγράμματα της Ένωσης. Τον Απρίλιο του 2012 οι αρχές της Αρμενίας συμμετείχαν, άρχισαν να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά της ΕΕ και των υπηρεσιών. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα. Δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει η Αρμενία σε προγράμματα επιστημονικά, έρευνας και τεχνολογικά προγράμματα και να προσεγγίσουν οι πολίτες ε, αυτής της χώρας ε, την ΕΕ. Όλα αυτά τίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής μας ε, για την γειτονία. Και Προφανώς γνωρίζετε ότι υπήρξαν σημαντικά συμβάντα σε, αυτή την, ε, σε αυτές τις εξελίξεις τα τελευταία, το τελευταίο διάστημα. Για να μας εισαγάγει τα θέματα αυτής της έκθεσης, ε, ο κύριος Πορέμπα δεν παρίσταται, αλλά ο κύριος Τάνοκ θα τον εκπροσωπήσει και έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, μιλώ εκπρόσω, ως εκπρόσωπος του συναδέλφου μου ε, που δεν μπορεί να έρθει εδώ γιατί είναι άρρωστος. Όλοι σκεφτόμαστε ακόμα την πρόσφατη απόφαση που δεν μας εξέπληξε του Προέδρου της Αρμενίας που θα ενταχθεί στην Ρωσική Τελωνιακή Ένωση. Ε, δεν είναι η καλύτερη ε, χρήση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, τις πρόσφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα, δεν θα συμμετάσχει η Αρμενία στην, ε, στις προσπάθειες αυτές. Ε, οι αρχές του Γέρεβαν είπαν ότι θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μεταρρυθμίσεις και τον εξυγχρονισμό της χώρας. Η σύσταση που συζητάμε σήμερα του κυρίου Περέβο, εκ μέρους της Επιτροπής μας, είναι τμήμα της στρατηγικής που ε, ξεκίνησε με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινωνία και απορρέει από μια απόφαση του Συμβουλίου του Μαρτίου του 2007 για τη δυνατότητα ε, οι χώρε αυτέ να συμμετέχουν πλήρω σε επιλεγμένα κοινοτικά προγράμματα και οργανισμού ω μέτρο ε, που σκοπό έχει την προώθηση του εξυγχρονισμού των μεταρρυθμίσεων και τη μετάβαση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ε, Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πολιτιστικέ εκπαιδευτικέ, ε, περιβαλλοντικές, τεχνικές επαφές, ε, επαφές μεταξύ ανθρώπων ε, και τομιακή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η διαδικασία είναι χωριστή από την Συμφωνία Συνεργασίας και έχει μονογραφηθεί ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η Συμφωνία Συνεργασίας θα συζητούνταν στο Βίλνιο στο Βίλνιους τον Νοέμβριο και θα μονογραφούνταν τότε, αλλά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλει ο εισηγητής να συνδεθεί αυτή η σύσταση με την πρόσφατη απόφαση που πήρε η αρμενική κυβέρνηση και που θα επικυρωθεί από ένα δημοψήφισμα ε, να, ενταχθεί στην, να στην ε, Τελωνιακή Ένωση της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ε, το να τη στρέψουμε την πλάτη τώρα θα είναι προς όφελος της Ρωσίας. Υπάρχουν νέε μορφέ συνεργασία και είμαστε έτοιμοι για νέε μορφέ συνεργασία με την Αρμενία, η οποία είναι ενεργό ε, εταίρο στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Συνεχίζει τι ε, μεταρρυθμίσει που τη πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τμήμα ακόμα τη κοινοβουλευτική συνέλευση. Γι' αυτό λοιπόν ο εισηγητή είπε να δώσουμε τη συνένεσή μας για μια συμφωνία πλαίσιο ε, με σκοπό τη συμμετοχή της Αρμενίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπάρχει και ένα επεξηγηματικό μνημόνιο στην σύσταση αυτή. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση δίνοντας τον λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Κουσμάτσεφ πρώτος, εξ ονόματος του ΕΛΚ παρακαλώ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τη γνώμη του εισηγητή. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε τις τελευταίες πολιτικές εξέλιξεις στην Αρμενία και την πίεση της Ρωσίας τώρα στην κυβέρνηση της χώρας αυτής να ενταχθεί στην Τελωνιακή Ένωση η δε σύσταση αφορούσε την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν πακέτο με μια άλλη ε, πρόταση την οποία έχουμε ήδη εγκρίνει για την επανεισδοχή και τις θεωρήσεις και δεν είναι άρα νομίζω καλό σημάδι να αρχίσουμε τώρα να στρέφουμε τα νότα μας στην Αρμενία και να δυσκολεύσουμε ακόμη περισσότερο την δύσκολη κατάσταση ε, που αντιμετωπίζει η Αρμενία. Στηρίζω λοιπόν την σύσταση του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λούνα Τσεκ παρακαλώ. Um, Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω πως σε γενικές γραμμές υποστηρίζουμε τη θέση του εισηγητή πως παρά την απόφαση του Πρόεδρου της Αρμενίας να ενταχθεί στην Ευρασιατική Τελωνιακή Ένωση θεωρούμε πως η συμμετοχή στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο βοηθάει τους πολίτες και τους ανθρώπους στην Αρμενία και όχι την κυβέρνηση τόσο. Γι' αυτό θέλουμε να τη στηρίξουμε αλλά έχουμε μια μεγάλη ανησυχία ε, που είναι ήδη το πρόβλημα που είχαμε και με την ε, διευκόλυνση βίζας. Το ότι δεν γίνεται δηλαδή διάκριση μεταξύ Αρμενίων πολιτών που κατοικούν στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και ήδη ε, με την διευκόλυνση βίζας το ρωτήσαμε Μα είπε η Κομισιόν πω δεν γίνεται καμία διάκριση αφορά του Αρμένιου πολίτε όπου και αν κατοικούν. Το πρόβλημα είναι πω αυτό σημαίνει πως όσοι δεν είναι Αρμένοι οι πολίτες και κατοικούν στον Αγκόνο Καραμπάχ δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ξέρουμε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η Αρμενία κατέχει το 20% της έκτασης του Αζερβαϊτζάν. Οπότε το ερώτημά μου είναι γιατί δεν είχαμε εξηγήσει κάτι ή γιατί συμπεριλήφθηκε κάτι στο επεξηγηματικό σημείωμα και το άλλο είναι τι γίνεται με τα προγράμματα της Ένωσης με το Αζερβαϊτζάν, γιατί η πρότασή μας είναι να ψηφίσουμε ταυτόχρονα τις ε, δύο συμφωνίες για ε, τις, ε, τις και το Αζερβαϊτζάν για να ισχύσει ταυτόχρονα γιατί έτσι ευνοείται οι Αρμενοί, ευνοούνται οι πολίτες της Αρμενίας και αυτοί που κατοικούν στον Αγκόνο Καραμπάχ που ξέρουμε ότι είναι κατεχόμενη περιοχή. Και πρέπει να είμαστε σαφείς. Όταν μιλάμε για τη Γεωργία, μιλάμε και για την ε, Απχαζία και την Νότια Οσετία, για τους πολίτες που έχουν ρωσικά διαβατήρια στις κατεχόμενες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφής η γραμμή μας και θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν πώς έχουν τα πράγματα με το Αζερβαϊτζάν και θα ήθελα να συζητήσω να συμπεριλάβουμε ένα επεξηγηματικό σημείωμα. Αλλιώς δεν είμαστε συνεπείς με τη θέση μας παρόλα αυτά ως πράσινοι θα το υποστηρίξουμε γιατί εμείς θέλουμε να μπορούν να λάβουν όλες τα προγράμματα της Ένωσης. Ευχαριστώ κύριος Μπάγκερ τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ φυσικά βλέπω όφελος προφανώς να μπορέσει η Αρμενία να συμμετάσχει στα προγράμματα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να πιέσουμε την Αρμενία και να την απομονώσουμε η χώρα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με γειτονικέ χώρες. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την Τουρκία, υπάρχει πρόβλημα με το Αζερβαϊτζάν και φυσικά έχουμε και το πρόβλημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του ορεινού Καραμπάχ. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε έτσι ελαφρά την καρδία να πούμε ότι η Αρμενία οδηγήθηκε και πιέστηκε στο να βρεθεί την αγκαλιά της Ρωσίας υπό τον έλεγχο της Ρωσίας για παράδειγμα έχοντας ε, ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ε, στην επικράτειά της και ουσιαστικά τροχοπεδώντας, παγώνοντας ε, το πρόβλημα στο ορεινό Καραμπάχ και θέτοντας επιπρόσθετη επιβάρυνση βάρος στις δυσκολίες που υπάρχουν για την επίλυση αυτού του προβλήματος ήδη δηλαδή για την αναζήτηση μιας λύσης σε αυτό το ακαθόδες πρόβλημα είναι λοιπόν <clears throat> καλό να μην συνδέσουμε αυτή τη στιγμή όλα αυτά και να ανοίξουμε την δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτά τα προγράμματα η Αρμενία. Από την άλλη όμως πλευρά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι δεν είμαστε εμείς οι ΕΕ που εμείς ε, επιθυμούμε να κλείσουμε ή θέλαμε να κλείσουμε την πόρτα όσον αφορά την ε, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Σύνδεσης ε, ήταν από πλευράς της Αρμενίας αυτό το οποίο έγινε και δεν ήταν μόνο κάποιες ε, δηλώσεις που έγιναν έτσι σε κάποιες εφημερίδες αλλά ήταν δεσμευτικές δηλώσεις του Προέδρου της ίδιας Αρμενίας να μην το αγνοούμε αυτό, να μην το αμελήσουμε και να μην θεωρείται η Αρμενία ότι είναι θύμα τρίτων χωρών θυματοποιήθηκε. Πρέπει να επομιστούν και τις δικές τους ευθύνες οι Αρμένοι. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Κυρίλοφ, παρακαλώ. Uh, thank you, Chair. <coughs> Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως θυμόμαστε, στην τελευταία ολομέλεια συζητήσαμε το θέμα και βεβαίως ασκήσαμε κριτική στη ρωσική πίεση. Αν και οι τελευταίες πληροφορίες μου λένε πως δεν ήταν τόσο μεγάλη πίεση. Η απόφαση λήφθη σχετικά εύκολα. Βέβαια συμφωνώ με τον εισηγητή πως δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να κλείσουμε την πόρτα εντελώς γιατί τότε θα δείξουμε πως κάνουμε και εμείς τα ίδια. Να ασκούμε και εμεί πίεση. Α αφήσουμε λοιπόν αυτή την πόρτα. Συμφωνούμε με τις δηλώσεις επίσης του Επιτροπού Φίλε στην επίσκεψή του στην Αρμενία. Και πρέπει να έχουμε κατά νου πως πολλοί αρμένοι πολίτες θα ικανοποιηθούν από την εξέλιξη των σχέσεων, τουλάχιστον όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, κάποια προγράμματα που αφορούν τους νέους, ανταλλαγές, εκπαίδευση κτλ. Θα τα δουν θετικά. Βεβαίω πρέπει να έχουμε και ένα νέο φόρουμ και πολιτικά νομίζω είναι σαφές πως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι τα πράγματα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Αλλά νομίζω πως μετά από την απόφαση αυτή πρέπει να συνεχίσουμε τις ανταλλαγές, τα προγράμματα και αυτό το οποίο έχει ζωτική σημασία είναι να ξεκινήσουμε να κινητοποιούμαστε στο θέμα του μεγόρνο Καραμπάχ. Αφορά ανθρώπους, αφορά εδάφη και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ε, δεχόμαστε το status quo και λέμε υποστηρίζουμε την ομάδα του Μίνσκ. Η ομάδα του Μίνσκ δεν έχει κάνει τίποτα 20 χρόνια και δεν υπάρχει πολιτική παρουσία αν δεν κάνουμε κάτι όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης. Το ίδιο και με τις άλλες συγκρούσεις του Νοτιού Καυκάσου, αλλά και στην υπερθυνιστερία. Και, μία που δεν κάναμε τίποτα για την επίλυση αυτών των παγωμένων συγκρούσεων, αλλά μετά ασκούμε κριτική. Ότι ασκείται πίεση στη χώρα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι πιο θετικό. Για να είμαστε σε διαφορετική κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι ευρωπαϊκό έδαφος αυτό. Είμαστε μια μεγάλη ένωση, πρέπει να έχουμε επιρροή, τουλάχιστον ιδέες. Δηλαδή, μία επίσκεψη της κάθε μας στην περιοχή δεν αρκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πέρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ διστακτικός απέναντι σε αυτή την πρόταση του εισηγητή που λέει ότι το ε, Κοινοβούλιο εγκρίνει την ε, σύναψη του πρωτοκόλλου. Εγώ έτσι πως καταλαβαίνω τα πράγματα, η Αρμενία έκανε μια εχθρική κίνηση. Γιατί ο Πούτιν δεν είναι φίλος μας. Και έκανε λοιπόν μια επιλογή. Είχε αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία καλύπτεται και από αυτό που συζητάμε σήμερα. Και την ένωση, ανάμεσα αυτό και στην ένωση με τον Πούτιν και τους κολλητούς του, οι οποίοι μας τραγουδούν τραγούδια εντελώς εχθρικά, καθόλου φιλικά, νομίζω ότι η επιλογή ήταν σαφής. Ίσως εντάξει, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να κλείσουμε εντελώ την πόρτα, αλλά ας την κρατήσουμε μισάνοιχτη, όχι ορθάνοιχτη. Αν πούμε ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλου, ανοίγουμε ορθάνοιχτη την πόρτα, αλλά και δεν συνέβη τίποτα. Εγώ νομίζω το πολιτικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε μετά από τις τελευταίες αποφάσεις του Αρμένιου Προέδρου είναι σαφές. Αυτή η σύνδεση, αυτή η συνεργασία με τον Πούτιν είναι μια μη φιλική χειρονομία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να ψηφίσω το κείμενο όπως έχει τώρα. Χρειάζεται κάτι καινούριο, γιατί είναι μια πολιτική χειρονομία που έκανε η Αρμενία, έτσι πρέπει να την ερμηνεύσουμε, αλλιώς δεν βοηθάμε τους Αρμένιους ε, πολίτες. Γιατί αν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με, την, ε, με αυτό το νέο ε, προσανατολισμό της Αρμενίας, με αυτή τη στροφή της Αρμενίας προς τον Πούτιν, τότε είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε εμά και στον Πούτιν. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πολιτική, στο πολιτικό όραμα του Πούτιν και στο πολιτικό όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Κυρία Λούνατσεκ. Δυστυχώς δεν υπάρχει εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κρίμα. Ο κύριος Βαλτζάν είναι εδώ. Δεν ξέρω αν άλλος θέλει. Κύριε Τάνο, θα σας ξαναδώσουμε το λόγο. Διαμαρτυρόμαστε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την κυρία Άστον. είναι καθοδόν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ώστε να μπορέσει όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθεί αυτό το θέμα να δώσει κάποιες απαντήσεις στις παρατηρήσεις. Έχει τον λόγο ο κύριος Μπατζανή και τελευταίο θα είναι ο κύριος Τάνοκ για να κλείσει η συζήτηση. Μπουλιάνιτς, περδόν. ζητώ συγγνώμη. Εδώ και καιρό προσπαθούμε να πείσουμε οι μεν τους δε Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για εχθρική στάση της Αρμενίας. Η χειρονομία του Αρμένιου Προέδρου ε, είναι αποτέλεσμα έντονων πιέσεων που του ασκήθηκαν από τους Ρώσους. Οι Αρμένοι κάναν μια αξιολόγηση και αποφάσισαν τι πρέπει να κάνουν. Τώρα, απόκειται σε εμά να πούμε ότι δεχόμαστε την απόφαση. Είναι δική τους απόφαση. Και έχουν δικαίωμα να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Φυσικά, έχουμε δύο ομάδες φίλων, ε, γειτόνων. εκείνοι που έχουν πιο έντονες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και θα προσπαθήσουν να γίνουν ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εγγύς μέλλον και εκείνοι που δεν έχουν τέτοιες φιλοδοξίες. Προφανώς οι Αρμένοι ανήκουν στη δεύτερη ομάδα γειτόνων αυτή τη στιγμή, προς το παρόν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε επικοινωνία, επαφή και καλές γειτονικές σχέσεις με αυτή τη δεύτερη ομάδα γειτόνων. Με αυτούς δηλαδή που δεν έχουν πια ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Υπό την, έννοια, υπό την έννοια των υπολείπων χωρών της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, Μολδαβία, Ουκρανία κτλ. Ακόμα και να έχουν αποφασίσει διαφορετικά, μπορούμε να έχουμε σχέση μαζί τους. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να διαμηνήσει ο εισηγητής. δεν μπορούμε και δεν θα μείνουμε αμέτωχοι. Μα είπε όχι για ένα είδος σχέσεων. Υπάρχουν άλλα είδη σχέσεων που μπορούμε να αναπτύξουμε και οι οποίες μπορεί να είναι επωφελείς και για μας και για την άλλη χώρα, ας πούμε, όπως η Αρμενία. Θα υπάρξουν και άλλες χώρες που θα βρεθούν σε αυτήν ε, θέση στο μέλλον. Δεν θα ήθελα να κάνουμε μια σκληρή κίνηση και αυτή η κίνηση να αποτελέσει προηγούμενο στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τάνοκ παρακαλώ. ναι, ναι, ναι κύριε Λούνατσεκ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να τοποθετηθώ πρόεδρε σε αυτό που είπατε για το ότι θα έρθει κάποιος λέει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας επεξηγήσει κάποια πράγματα. Δύο εδώ έχω. Ναι, όταν εκείνος ή εκείνη έρθει. Αλλά ήδη είχαμε μια δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το αίτημα συναδέφου για τις θεωρήσεις διαβατηρίων, visa facilitation, θα ήθελα να μην μας δώσουν την ίδια απάντηση όπως τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν είπαν τίποτα τότε σχετικά. Επίσης και για τον κύριο Τάνοκ που εκπροσωπεί τον ε, εισηγητή κύριο Πορέμπα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να πείτε στον κύριο Πορέμπα αυτό. Θα ήταν σκόπιμο για την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αιτιολογική σκέψη, ε, στις αιτιολογικές ε, να εκφράσουμε την ανησυχία μας για πολίτες ε, ή όσους ζουν στον Αγκόρνο Καραμπάχα και να αναφέρω ότι εσείς είσαστε εκείνος που ανέφερε το θέμα των ε, υπηκών με ρωσικά διαβατήρια και σε σχέση και με την Απχαζία. Θα πρέπει το ίδιο να πούμε όταν ε, έρχεται η ώρα να εξετάσουμε τα θέματα του ορεινού Καραμπάχα και να δούμε ότι αυτό θα πρέπει να διαβιβαστεί στον κύριο Πορέμπα να τα εντάξει αυτά στις αιτιολογικές σκέψεις. Την ανησυχία μας για την κατάσταση αυτών των ανθρώπων εκεί. Σας ευχαριστούμε κύριε Αλούνα. ο κύριο Τάνοκ. Χαίρομαι για το έτοιμά σας, εγώ δεν θα το υποστήριζα. Ε, είμαι φίλος της Αρμενίας και για να είμαι ειλικρινής η ερμηνεία που κάνετε του διεθνούς δικαίου δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία έχει πει το Κοινοβούλιο για το θέμα του Ναγκόρνο Καρμπάχ. Εμεί λέμε πως το Ναγκόρνο Καρμπάχ είναι σε μία αμφισημία κάπου μεταξύ αυτοδιάθεσης ε, ή εδαφικής ακεραιότητας ε, του Αζερβαϊτζάν. Δεν, αναλόγως με το τι θα γίνει στη διαδικασία του Μίνσκ. Οι δε περιοχές γύρω από τον Αγκόρνο Καραμπάχα δεν κατοικούνται πλην του στρατού. Δεν έχω πάει βέβαια στο ίδιο τον Αγκόρνο Καραμπάχ παρά μόνο στο Αζερβαϊτζάν. Από όσο ξέρω δεν υπάρχουν εκεί πέρα μη Αρμένοι Οπότε αυτά τα οποία λέτε περί μία Αρμενία δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά τέλος πάντων είναι λίγο ακαδημαϊκό το ζήτημα. Δεδομένη στις θέσει που πάντα είχαμε σε σχέση με την ομάδα του Μίνσκ, οπότε εγώ δεν θα έλεγα στον Τόμας να υιοθετήσει την θέση σας. Μπορείτε να υποβάλλετε βεβαίως τροπολογίες και να ψηφιστούν. Για τα σχόλια του κυρίου Πρέντα δεν συμφωνώ μαζί του. Ε, έχει μια σοβιετική άποψη όπου ένας κερδίζει κάτι που χάνει ο άλλος. Προσφάτως η Ισλανδία ε, αρνήθηκε να ενταχθεί και θεωρήθηκε κάτι το εχθρικό, ότι ήθελαν απλά να μπουν στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. με είναι δικαίωμά του. Το ίδιο και της Αρμενίας. Ε, Δυστυχώ βεβαίω στράφηκε στην Ρωσία γιατί είναι η μόνη στρατιωτική εγγύηση που έχει όσον αφορά την κυριαρχία της θα ήταν δύσκολη απόφαση και είμαι σίγουρος πως ασκήθηκε κάποια πίεση δεδομένου του ότι η Ρωσία είχε υποσχεθεί λίγο πολύ να πουλήσει ένα δισεκατομμύριο όπλα στον Πακού. Αλλά φίλος της Ρωσίας δεν σημαίνει εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν είναι σωστό αυτό και πρέπει να αφήσουμε νομίζω ανοιχτή την πόρτα ε, προς την Αρμενία γνωρίζοντας πως ε, έχουν κάνει μια στρατηγική επιλογή, αλλά βέβαια τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον, οπότε το να κλείσουμε τώρα αυτή την πόρτα θα ήταν λάθος. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Λούνατσεκ. Ξανά. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω, ε, είπατε πως είστε φίλος Αρμενίας, μα δεν είναι θέμα φιλίας, είναι θέμα αρχής. και ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Οπότε θα ήθελα, εγώ θα ζητήσω από τους υπόλοιπους και να συντάξω μια γνωμοδότηση. Από όσο ξέρω δεν μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις σε επεξηγηματικές δηλώσεις. Οπότε θα ζητήσω, θα ρωτήσω τους, ε, θα ρωτήσω τους εάν μπορούμε να κάνουμε μια ε, αφεξηγηματική δήλωση. Επίσης, όπως ακούσατε, και η ομάδα μου υποστηρίζει τη συμμετοχή της Αρμενίας σε προγράμματα της Ένωσης. Δεν θα το καταψηφίσουμε. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, δεν έχει λυθεί. Οπότε η ανησυχία μας πρέπει να είναι, πρέπει να αναφερθεί στη δήλωση. Θα ρωτήσω εγώ λοιπόν τους κοιόδες ε, εάν μπορούν να υποστηρίξουν ε, αυτό το οποίο θέλω να κάνω σε σχέση με τον κύριο Πορέτα. Ε, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση λοιπόν για αυτό το θέμα. Σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών εκπνέει στις 25 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι 12.00. Και τώρα θα κλείσει η συνεδρίασή μας για 8 λεπτά για να μπορέσουμε να ακούσουμε τη δήλωση που θα κάνει ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιγυρία και κλεισμένων των θυρών, η κυρία Λούνατσεκ. Μόλις είπατε ότι υπάρχουν τροπολογίες που θα κατατεθούν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Μόλις σας είπα δεν υπάρχουν τροπολογίες, δεν υπάρχουν τροπολογίες από ό,τι κατάλαβα. Όχι, πιστεύω ότι η ερμηνεία που η γραμματεία έδωσε ήταν αν θα μπορούσαν να κατατεθούν τροπολογίες ε, στο, στις αιτιολογικές σκέψεις. Αυτό είναι υπό τη διακριτική ευχέρεια του εισηγητή. Εν πάση περιπτώσει η κατάθεση τροπολογιών στο κείμενο από πλευρά του νόμιμου κειμένου από πλευρά των μελών της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής αυτή η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών εκπνέει στις 25 Σεπτεμβρίου στις 12 θα διακόψουμε για λίγα λεπτά ή 8 λεπτά ώστε στις 5 να αρχίσουμε με την ε, έκθεση των ε, παρατηρήσεων του επικεφαλής αντιπροσωπή.